Θέλουμε να διασφαλίσουμε την αγορά εργασίας και να διασφαλίσουμε το δικαίωμα στην απεργία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Εξ ονόματος της Επιτροπής θα λάβει το λόγο ο Αντιπρόεδρος, ο κύριος Σιμ Κάλλας. Έχετε το λόγο κύριε Κάλλας